τον εισηγητή και πρόεδρο της ε, Ομάδας Εργασίας για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Σταδιακής και Πολιτικής Ανάλυσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Έληξε η συζήτηση για αυτό το θέμα. Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα γίνει η ψηφοφορία. Και τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι η έκθεση Ρέγνερ. Το λόγο έχει η κυρία Εβελίν Ρέγνερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Επίτροπε, δεν έχει περάσει πολύ καιρό από τότε που εδώ στο Κοινοβούλιο ασχοληθήκαμε με τον κανισμό Βρυξέλλες 1. Και όχι μόνο ασχοληθήκαμε με τον κανονισμό αυτό, αλλά ως Ευρωπαίοι νομοθέτες ε, συμμετείχαμε επικοδομητικά στην αναδιατύπωση του κανονισμού. Από το 2012, από το Δεκέμβρη συγκεκριμένα, υπάρχει μια νέα διατύπωση για τη δικαστική αρμοδιότητα και την εκτέλεση αποφάσεων σε θέματα εμπορικά και αστικά. Ε, υπάρχουν πάρα πολλές βελτιώσεις, γιατί εδώ αδιαμφισβήτητα πρόκειται για υπεραξία που προσφέρεται στους ε, πολίτες ε, τους, της Ευρώπης κάποιες διαδικασίες προβλεπόντουσαν καταργήθηκαν και στο μέλλον θα είναι πολύ πιο εύκολο ε, να γίνονται εκτελεστές οι πράξεις. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στην ε, διαδικασία αυτή, η επέλεξη στη διαδικασία αυτή την αναπομπή και γι' αυτό ε, αφαίρεσε κάποια στοιχεία που κατά τη δική μου όμως άποψη και της Νομικής Επιτροπής είναι πολύ σημαντικά. Συγκεκριμένα η διαδικασία καλύπτει ε, κάποια στοιχεία αλλά αφήνει πάρα πολλά άλλα. Η, σύνδεση ανάμεσα στην αρμοδιότητα για εργασιακά θέματα και ε, την αρμοδιότητα για την σύνταξη των, ε, και σύσταση των εργασιακών συμβολών δεν λαμβάνεται υπόψη. Μην ξεχνάτε όμως ότι ο εργασιακός βίος έγινε διασυνοριακός. Αυτό φαίνεται σε διάφορες αποφάσεις, Τόρλαν και Βάκινγκ, παραδείγματος χάρη, που κατά την άποψή μου πρέπει να αντιδράσουμε πρέπει εδώ ε, κάτι να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή η έκθεση βασίζεται στην αρχή ότι οι υπάρχουσες εργασιακές διατάξεις των κρατών μελών λόγω των ε, ε, αποφάσεων άλλων δικαστηρίων υπονομεύονται και πρέπει να προστατευτούν. γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πούμε ότι αρμόδια είναι τα δικαστήρια εκείνα όπου ισχύει και το εργασιακό δίκαιο. Θα πρέπει λοιπόν να ισχύουν όπως είπα οι αποφάσεις του κράτους που ε, λαμβάνει η χώρα η όλη υπόθεση. Αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να ισχύει για όλα τα εργατικά θέματα και για τις εργασιακές συμβάσεις η έκθεση ασχολείται με κάτι που είναι πολύ σημαντικό σε διεθνές επίπεδο, την αδύναμη πλευρά. Και στην αδύναμη πλευρά πολλές φορές ανήκουν άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται και εμπλέκονται σε εργασιακές αντιπαραθέσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η Κομισιόν στο μέλλον θα πρέπει να μελετά εντελεχέστερα τα θέματα τα εργασιακά και όχι να καταφεύγει μέσω στην αναπομπή τα εργασιακά θέματα ε, αφορούν τα συνδικάτα. Βεβαίως υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με τη χώρα, αυτό που ενδεχομένως προστατεύεται στη μία χώρα, σε μία άλλη χώρα δεν ισχύει και μπορεί να είναι και παράνομο. Γι' αυτό λοιπόν εγώ προτείνω η διατάξη του κανονισμού Βρυξέλλες 1 και με τον επόμενο κανονισμό ε, θα πρέπει να ταυτίζονται με τις διατάξεις που ισχύουν ε, για την υπετιότητα οι διατάξεις ε, περί μέσων ε, εργατικών αγώνων ε, θα πρέπει να ισχύουν για το κράτος όπου γίνονται οι αγώνες αυτοί. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσέξει τα θέματα αυτά. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μεμονωμένες επιχειρησιακές συμβάσεις θα πρέπει να επιδεικνύει μεγαλύτερη προσοχή. Ο κανονισμός Βρυξέλλες 1 ήδη περιλαμβάνει τώρα προστατευτικές διατάξεις για τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές. Ε, το κριτήριο ε, της, ε, του χώρου εγκατάστασης όπου έχει εγκατασταθεί ο εργαζόμενος, αυτό πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα κυρίως στις μεταφορές. Προφανώς δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στην εγκατάσταση και στον χώρο εργασίας. Μια επιχείρηση μπορεί να έχει εγκατασταθεί σε μια χώρα και τα μέσα μεταφοράς να έχουν καταγραφεί σε άλλη χώρα. Τότε λοιπόν μπορεί και το management και ο εργαζόμενος να βρίσκονται σε πάλι τρίτη χώρα. Βλέπετε λοιπόν ότι πρόκειται για περιπτώσεις που υπάρχουν και που απαιτούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να προσέξει τα θέματα αυτά περισσότερο, κυρίως ε, την αρχή της προστασίας ε, του αδυνάμου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω κανέναν που έχει ζητήσει κάτι the Εντείνω λοιπόν το λόγο στην κυρία Μαρία Δαμανάκη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Επιτροπή ευχαριστεί τον την εισηγήτρια, την κυρία Ρέγνερ και το Κοινοβούλιο που θέτει το θέμα της ε, δικαιοδοσίας σε θέματα εργασιακά. Ε, ε, συμμεριζόμαστε το στόχο της διασφάλισης της σωστής ε, προάσπισης των δικαιωμάτων των ανθρώπων που εργάζονται, αλλά και αυτών που κάνουν εργασιακούς αγώνες γενικότερα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ενισχυθεί, ότι έχει ενισχυθεί και θα πρέπει να ενισχυθεί στην νέα διατύπωση του κανονισμού Βρυξέλλες ένα αυτό το δικαίωμα ε, θα πρέπει να δοθεί το δικαίωμα στους ε, απασχολουμένους να έχουν ε, πρόσβαση στα ευρωπαϊκά δικαστήρια ακόμα και αν ο εργοδότης είναι εκτός Ευρώπης. Η Κομισιόν θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των νέων κανόνων τα επόμενα χρόνια. Θα δώσει μεγάλη προσοχή στην διαδικασία των ε, θεμάτων αποσχόληση που θέτει το Κοινοβούλιο. Αυτό μπορούμε να το εξετάσουμε μέσα στα πλαίσια τη αναθεώρηση που βλέπετε ε, στο άρθρο 79 του κανονισμού για την αναδιατύπωση. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η Κομισιόν στο μέλλον θα εξετάζει το ζήτημα των εργασιακών συμβάσεων. Αυτό μπορεί να γίνει εξετάζοντας πιο συγκεκριμένα την ε, ρήτρα αναδίπλωσης του άρθρου 21 σε υποθέσεις ε, εργοζομένων κατά εργοδοτών ε, στην ε, διατύπωση ενός πλαισίου όπου ο απασχολούμενος έχει, λαμβάνει οδηγίες σε καθημερινή βάση και αυτό γίνεται στον χώρο που δουλεύει και όχι εκεί όπου είναι η... ο εργοδότης. Ευχαριστούμε πολύ. Κλείνει η συζήτηση στην έκθεση Φράγα Εστέβες και δίνω το λόγο στην κυρία Φράγα Εστέβες.